Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο θα εκφράσει τη θέση του όσον αφορά την πρόταση ευθυγράμμισης ε, του ε, κανονισμού ε, ελέγχου της τήρησης με την συνθήκη της Λισαβόνας. Το Κοινοβούλιο είναι θεματοφύλακας της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Την πρόταση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ε, λαμβάνει υπόψη είναι τις παλιές αρμοδιότητες της επιτροπολογίας βάζοντάς τες είτε σε κατεξουσιοδότηση είτε σε εκτελεστικές πράξεις. Βεβαίως πέρα από το τυπικό του πράγματος θα πρέπει να μελετήσουμε τα κριτήρια κατανομής τα οποία βεβαίως ορίζονται από τη συνθήκη αλλά στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε μία θεά ζώνη συχνά ε, ε, εσφαλμένα ε, ξεχνούμε, λησμονούμε ότι η διαδικασία της, των αρμοδιοτήτων μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας χρειάζεται ευθυγράμμιση η οποία όμως θα πρέπει να γίνει με πολύ σωστό τρόπο. Κατεξουσιοδότηση πράξης λοιπόν οι οποίες εκ των υστέρων θα επιβεβαιώνουν από το Κοινοβούλιο το οποίο όμως είναι υπεύθυνο υπεύθυνο για αυτές. Ε, επομένως θα πρέπει να προσέχουμε ε, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τους πόρους τεχνικούς και ανθρώπινους για να κάνει αυτόν τον εκ των έλεγχο. Με τον ίδιο τρόπο ε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Κομισιόν στην γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας. Η ευθυγράμμιση με την Συνθήκη Λειτουργίας της Λισαβόνας βεβαίως θα πρέπει να γίνει ωστόσο τα άρθρα 290 και 291 ε, που ε, αφορούν την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως παράρτημα της συνθήκης δεν πρέπει να παραβλεφθούν. Η νομική επαλήθευση έχει γίνει λοιπόν όσον αφορά τον κανονισμό ελέγχου της ε, ε, αλίας. Πρέπει να πω το εξής. Ε, σωστή και συνεκτική εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν θα έλεγα ότι πρέπει να προωθήσουμε την κατεξουσιοδότηση πράξης έτσι ώστε οι αλίες οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Κατά δεύτερον λόγο, ε, ακολούθησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όταν αναφέρεται στην νομική ευθυγράμμιση ε, και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή και αναθεώρηση του, της, του κανονισμού για την αλλιευτική πολιτική παρά τις πολλές τροπολογίες ε, εγώ ε, αποφάσισα ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να λάβει υπόψη στον νέο κανονισμό για τον έλεγχο της αλληλείας της τροπολογίας. Γι' αυτό λυπάμαι πραγματικά πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέρχεται με μια πρόταση η οποία δεν έλαβε καθόλου υπόψη όλες αυτές τις προτάσεις. Στην ουσία μας έχει δώσει η Κομισιόν ένα κείμενο omnibus το οποίο δεν ελαμβάνει υπόψη καθόλου τις δικές μας απόψεις όσον αφορά την κοινή ελιευτική πολιτική ε, και τις απόψεις μας σχετικά με την ευφυή ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο της μεταρρύθμισης ε, και τις παρατηρήσεις ε, των συναδέλφων που γνωρίζουν επιτόπου και εν της πράγμαση το τι κάνουν και τι ζουν οι αλληλείς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο έλεγχος είναι ενιαίος και δεν πρέπει να κατακαιρματίζεται. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να δεχόμαστε όταν μας πιέζουν για να νομοθετήσουμε στα γρήγορα. Η Κομισιόν θα πρέπει να ξανασκεφτεί λίγο την πρότασή της. Παρόλα αυτά, εγώ θα πρέπει, δηλώνω ότι θα παραμείνω προσκολλημένη στην αρχική δέσμευση που είχα αναλάβει. Η κυρία Επίτροπος Δαμανάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη προς την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ευθυγραμμίζει τον κανόνα για τους ελέγχους με τη συνθήκη της Λισαβόνα. Θα ήθελα όλος ιδιαίτερος να ευχαριστήσω την κυρία Τωμά, την εισηγήτρια, για τις προσπάθειες που έκανε για τόσο σημαντικό ζήτημα. Έχουμε λοιπόν μια νέα νομοθεσία που διέπει την κοινή αλλιευτική πολιτική, όπως μας είπε η κυρία Τομά. Και ναι, αυτή η νέα νομοθεσία ετέθησε ισχύ από την 1η ε, Πρώτη του 2014. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα καταλήξαμε σε μια πολιτική συμφωνία για τους νέους κανόνες χρηματοδότησης και προσβλέπω με ανυπομονησία στην επίσημη έγκριση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ε, αυτή τη συνενετική λύση, το αχύτερο δυνατόν. Φυσικά αναφέρομαι σε αυτή τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση, διότι θέλω να τονίσω πω αυτό το πλαίσιο είναι απολύτω απαραίτητο για μια αποτελεσματική εφαρμογή και για αποτελεσματικούς ελέγχους. Με τους νέους κανόνες ε, θα αποκομίσουμε τα ωφέλη για τις παράκτιες κοινότητες, ε, για τους αλείς και για τα αποθέματα μόνο αν επέλθει συμφωνία και εφαρμοστεί σωστά. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για μένα αλλά και για τον διαδοχό μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με την κυρία Τόμα ότι πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού περί ελέγχων αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η εφαρμογή γίνεται με συνέπεια και εξασφαλίζεται έτσι ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποσυζήτηση πρόταση αποσκοπεί ακριβώς το, στην κατοχήρωση τη δυνατότητας που θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή εκλεστικών και κατεξουσιδιώτηση πράξεων και ότι αυτό θα γίνει ε, βάσει των κανόνων της συνθήκης Λισαβόνας. Αυτό συζητούμε τώρα, συζητούμε εάν οι εκτελεστικές πράξεις και οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση συνάδουν με τη συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς γι' αυτό αποφαίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα σεβαστούμε απολύτως τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, δεν συζητούμε τροποποιήσεις ουσίας, συζητούμε μόνο την ευθυγράμμιση του συστήματος με την συνθήκη. Έτσι θα πρέπει να ερμηνευτεί η σημερινή συζήτηση. Από ό,τι κατάλαβα επίσης ε, έχουν ζητήσει κάποιοι βουλευτές του Κοινοβουλίου πλήρη αναθεώρηση του κανονισμού περί ελέγχων. Θα ήθελα όμως να σας ε, ε, να υπογραμμίσω συγγνώμη ότι αυτός ο κανονισμός εδέθησε ισχύ το 2010 και αυτή η εφαρμογή άρχισε από το 2011, οπότε ο κανονισμός αυτός έχει μια ιστορία μόνο δύο ετών, σας διαβεβαιώ ότι η λειτουργία των κανόνων μας ε, θα αποτιμηθεί εν ευθέτω χρόνο. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση. Πολύ συγκεκριμένα θα αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού της κοινής ελευτικής πολιτικής για τους ελέγχους κάθε πέντε χρόνια και ήδη αναφερόμαστε σε αυτό μέσα στον κανονισμό. Άρα μπορείτε να περιμένετε κατά το πρώτο ήμιση του 2015 την πρώτη έκθεση από πλευρά ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπής. Ε, αυτό συνιστά υποχρέωση για την Επιτροπή και ε, είναι η πρόθεσή μας. Οπότε ο κανονισμός Omnibus, ε, στον οποίο αναφερθήκατε, είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται εδώ. Έχουμε αρχίσει την προετοιμασία αυτού του κανονισμού και περιμένουμε την έγκριση της κοινή ελευτικής πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να απευθυνθούμε, δεν μπορούσαμε να απευθυνθούμε μάλλον νωρίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμέναμε την έγκριση λοιπόν. Μόλις έχουμε ε, αυτή την ε, έκθεση, την αξιολόγηση, θα κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ε, να αναθεωρήσει και πάλι ε, την ε, κοινή αλλιευτική πολιτική. Θα πρέπει Να διακόψω εδώ. Ε, έχω την εντύπωση ότι ε, στις αρχές ε, του 2015 ο διάδοχός μου θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, το δικό μας έργο μέχρι την εκπνοή της θητείας μας η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να εφαρμοστεί σωστά ο κανονισμός για τους ελέγχους και να γίνει αξιολόγηση στις αρχές του 2015 όπως προβλέπετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο. Δίνω τον λόγο στη συνάδελφο Φράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μου υποστηρίζει αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, θέλησή της να αποδεχθεί τις ε, προτάσεις μας που μας ε, επίτρεψαν να αντιμετωπίσουμε το θέμα της επιτροπολογίας. Ταυτόχρονα πιστώ... Μια αναθεώρηση του ελεγκτικού κανονισμού η νέα αλληλευτική πολιτική έχει σαν στόχο να μην βρεθούμε σε μια σειρά αλλαγών που θα υπόκεινται σε διάφορες ερμηνείες και θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε επιτάπητος, όπως ανέφεραν οι τρεις ε, προλαλήσαντες, την πρόταση Omnibus για να προσαρμόσουμε τις διατάξεις της νέας κοινή ελευτικής πολιτική στην απαγόρευση των απορρίψεων που περιλαμβάνει πάνω από 30 αλλαγές στην προγενέστερη εκδοχή του ελεγκτικού αυτού κανονισμού. Για το λόγο αυτό θα ήταν ευκταίο σε ένα κοντινό μέλλον εσείς ή ο επόμενος Επίτροπος να επανεξετάσετε διεξοδικά τον κανονισμό. Η δεύτερη σκέψη που προκύπτει από την ε, έκθεση αυτή είναι η ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση των της υπράξεων. Εγώ θέλω πάνω από όλου να έχουν εξουσίε στο Κοινοβούλιο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, το λέω αυτό για να το σκεφτούμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να εξετάσουμε μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει το Κοινοβούλιο στην ε, ελεγκτική δραστηριότητά του, ιδιαίτερα σε επιτροπέ με λίγα μέσα και λίγα μέλη. Το να μπούμε σε μια θεσμική υποχρέωση που δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τέλει με τις απαραίτητες εγγύησεις μπορεί να οδηγήσει σε αντιστροφή του νομίσματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η συνάδελφος ε, Ρόντες. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, από τη δική μου πλευρά νομίζω ότι υπάρχουν δύο βασικά κεντρικά ζητήματα στην πολιτική αλίας. Καταρχάς, ε, οι τα βιώσιμα αλλιεύματα, οι ποσότητες ε, αλλιευμάτων, οι, οι οποίες πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την κοινή αλλιευτική πολιτική. Ύστερα, η, τη μορφή της πολιτικής αυτήν την έχουμε ρυθμίσει στα βασικά της στοιχεία. Ε, στην, στο μέλλον θέλουμε να έχουμε περισσότερα ψάρια στην Ευρώπη. Ε, υπάρχουν κάποιοι, κάποιες βασικές αρχές ελέγχου που έχουμε θεσπίσει. Να είναι δηλαδή αποτελεσματικός, συντονισμένος και ανάλογος των συνθήκων ο έλεγχος. Ε, οι λεπτομέρειες δεν είναι οι κανόνες, ανήκουν στον ε, κανονισμό για τον έλεγχο. Ο κανονισμός για τον όλεγχο, τον οποίο προσαρμόζουμε στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας ε, σήμερα, είναι κάτι που πρέπει να γίνει, γιατί λίγο γιατί πρέπει οι Υπουργοί να ψηφίσουν αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, κατά την άποψή μου, ο όλεγχος ε, της αλληλεία στην Ευρώπη θα βελτιωθεί με αυτόν τον τρόπο. Παρ' αυτά με τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, και με την απαγόρευση της ε, ρήψη των αλλιευμάτων θα έχουμε τη δυνατότητα της απόρριψης των αλλιευμάτων θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πιο απλούς κανόνες. Μπορούμε για παράδειγμα σε πολλές περιπτώσεις να έχουμε ελάχιστα μήκη τα οποία καταργούνται. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόλις αποσφαλίσουμε ότι οι αλληλείς τηρούν τις απαγορεύσεις. Αλλιώς είναι αντιπαραγωγικό το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό λοιπόν ζητώ από την ε, ε, Κομισιόν να καταθέσει όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα νέο κανονισμό για τον έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ε, ο μελητής ο κύριος Νέλης. Ο Τόρβαλτ ε, αγαπητέ Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Ιζαμπέλ Τωμά και την Κάρμεν Φράγκα, την ε, σκιώδη εισηγήτρια, για τη συνεργασία που είχαν για τα τεχνικά ζητήματα του οργανισμού περιελέγχων τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Η αναθεώρηση κοινή αλληλευτική πολιτική που ανέκρινε πέρυσι το Κοινοβούλιο ε, σημείωσε μεγάλη πρόοδο σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη και τα βιώσιμα αποθέματα. Έτσι μπορούμε να διακόψουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο στον οποίο είχαμε έλθει την τελευταία δεκαετία. Αυτό σήμανε μειωμένα αποθέματα, μειωμένη βιοπικιλότητα και λιγότερες ε, θέσεις εργασίας. Ε, η μεταρρύθμιση ε, για να σημάνει πραγματική πρόοδο πρέπει να ακολουθήσει μια ορθή εφαρμογή. Η έλεγχη είναι βασικότατο εργαλείο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί στην πράξη η μεταρρύθμιση για να προστατεύσουμε τα αποθέματα, να προστατεύσουμε το περιβάλλον ε, και για να κρατήσουν ομοιόμορφες ε, συνθήκες ε, σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να εφαρμοστούν σωστά οι έλεγχοι και να καταπολεμηθεί η απάτη. Ε, με την σύσταση του Ευρωπαϊκού Αλλιευτικού Ταμείου ε, και την έγκριση των αυξημένων κονδυλίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό το ταμείο έχουμε ήδη καλύτερες ε, συνθήκες υπό τις οποίες θα εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη οι έλεγχοι. Έχουμε λοιπόν αυξημένα κονδύλια και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να έχει περισσότερες απαιτήσει από τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τα υπεσχημένα με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε βελτιωμένα αποθέματα, ε, καλύτερες ε, προοπτικές απασχόλησης για τις παράκτιες ε, κοινότητες και επίσης δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον αλληλευτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. και σας ευχαριστούμε για την ανεξάρτητη, αμερόληπτη και σοβαρή δουλειά που κάνατε στα πλαίσια της έρευνας για την Τρόικα. Ο κύριος Δρομέδα είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ε, επειδή έχω λίγο χρόνο θέλω να σταθώ στα βασικά. Ω εισηγητή για τον κανονισμό ελέγχου στην περασμένη θητεία, διαπίστωσα πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση των κανόνων. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να ενισχύσουμε. Αυτό είναι που πρέπει να εξασφαλίσουμε κατά βάση. Και με φοβίζει κάποιες τροπολογίες ε, που έχουν υποβληθεί αποδυναμώνουν το πλαίσιο και τον κανονισμό ελέγχου. Γι' αυτό θέλω να είμαι σαφής όταν θυμίζουμε αυτή τη στιγμή όχι μόνο την εντολή της μεταρρύθμισης της κοινή ελευτικής πολιτικής αλλά και το ότι ήδη πετύχαμε ως κοινοβούλιο να αυξηθεί ο προπολογισμό και για τον έλεγχο και για τη συλλογή δεδομένων να περάσει το κοινοβούλιο ένα σαφές μήνυμα ότι αυτό θέλουμε διότι αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι να αυτό που φοβάμαι είναι μήπως με αυτά που ψηφίζουμε περνάμε το ακριβώς ανάποδο μήνυμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόμπατσεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κοινή αλληλευτική πολιτική και, κανονισμοί και ο κανονισμός ελέγχου είναι βασική προϋπόθεση για να ελοποιηθεί η νέα ΚΑΠ. Η παρούσα φάση είναι καθοριστική για να προσαρμοστεί ο κανονισμός στις νέες απαιτήσεις της συνθήκης της Λισαβόνας ο στόχος της δουλειάς μας θα πρέπει να είναι να υπάρχουν οι, αναγκαίοι κανονισμοί για να μπορέσουν να γίνει σεβαστή η κοινή αλληλευτική πολιτική και όλες τις χώρες της Ένωσης με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν υπάρξει ενιαία, αν δεν υπάρξουν ενιαίες λύσεις δεν θα υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα όλων είναι ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν υπάρχουν στην πράξη. Άρα πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση τώρα. Ε, στην Βαλτική, για παράδειγμα, ε, και αλλού θα πρέπει να δούμε πόσο σημαντικό επιπτώσεις έχουν τυχόν λάθη της κοινή ελληνική πολιτικής. Μπορεί να προκύψουν προβλήματα και στον πληθυσμό του, του Μπακαγιάρου και στις ε, λειτουργίες της κοινή ελευτικής πολιτικής βλέπουμε ε, ότι σε περίπτωση που ο μπακαλιάρος δεν αλλιεύεται σωστά, μεγάλο κομμάτι του, ε, του ψαριού δεν μπορεί να πολυθεί ή χρησιμοποιείται για ηχθιάλευρα. Άλλα ψάρια, η ρέγγα για παράδειγμα, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Λοιπόν, ζητώ από εσά κύριε Επίτροπε να προσπαθήσετε να σταματήσετε τα προβλήματα που έχουμε στη Βαλτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ζωάν Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εν γέννη συμφωνούμε με τις προτάσεις της ηγήτριας, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα για το οποίο θέλουμε να επιμείνουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα ουσία όταν μιλάμε για του κανονισμού ελέγχου ε, ω προ την ορθή εφαρμογή του νέου κανονισμού τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Το πρόβλημα είναι οι κανόνε τη κοινή νέα ε, αλληλευτική πολιτική, διότι είναι κεντρική διαχείριση αποκομμένη από την πραγματικότητα ε, που δεν λαμβάνει υπόψη τη ιδιαιτερότητα κάθε περιοχή, του κάθε αλλιεύματο ε, και γι' αυτό έχουμε ε, καθιευθυντρίε γραμμέ ε, που είναι εντελώ ξεκομμένε Επομένω, από την πραγματικότητα που δεν προσαρμόζονται στον κάθε κλάδο και τελικά δεν εφαρμόζονται ή όταν εφαρμόζονται έχουν αντίθετα αποτελέσματα σε σχέση με τα αναμενόμενα. Και γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν ανάντι να ασχοληθούμε με τον έλεγχο για να τον διευκολύνουμε, διευκολύνοντας σε μία ε, εκ του σύνεγγης διαχείριση, προαγάγοντας την ευημερία του τομέα, όχι μόνο ως προς την εκτέλεση, αλλά ως προς την πραγματική οικονομική ζωή, εφαρμόζοντας την βασική αρχή της συνδυασμού Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μιλάν Ακούιντο Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια με την οποία συμφωνώ σχεδόν απόλυτα για το κείμενο που είπε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα στην επόμενη περίοδο να μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, νωρίτερα, διότι και ο κανονισμό ελέγχου έχει ένα βασικό πρόβλημα, χωρί συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Το είδαμε ε, ε, μετά την συναπόφαση, μετά τη συνδίκη τη Λισαβόνα, αλλά χωρί συναπόφαση. Ο κανονισμό δεν είναι εφαρμόσιμο. Το πρόβλημα εφαρμογή οφείλεται στο ότι ο κανονισμό έχει γίνει λάθο. Άρα πρέπει να αναθεωρηθεί ε, επιγόντως και εύχομαι ότι η πρόθεσή σας να προχωρήσετε γρήγορα σε έναν νέο κανονισμό ελέγχου να αποτελέσει στο, ε, καλή, ε, καλή προσέγγιση και να επιτρέψει να παρέμβει το Κοινοβούλιο στην διαδικασία αυτή. Να σας πω ότι είστε κάπως αισιόδοξοι, υπερβολικά, υπερβολικά αισιόδοξοι. Η πολιτική συμφωνία προδόθηκε από μια τεχνική συμφωνία που άλλαξε ουσιαστικά βασικά πολιτικά δεδομένα. Δεν είναι δεδομένο λοιπόν, τουλάχιστον η στάση της, η δεδομένη, τουλάχιστον η στάση της ομάδας μου για την σύναψη της συμφωνίας που αναφέρεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο. Ε, ε, ε, Πρόεδρε, να συγχαρώ και εγώ την εισηγήτρια να τονίσω ότι ο κανονισμός ελέγχου ήταν ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότητα της ελεκτικής πολιτικής με, 20, με ημερομηνία 20 ε, Νοεμβρίου του 2009, λίγες μέρες μετά τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, άρα πρέπει να, προβλεφ, να προσαρμοστούν οι ερμοδιότητες και τα, το περιεχόμενο του κανονισμού στις ε, κατεξοδότητες πράξεις που απαιτεί η Λισαβόνα. Ευχαριστώ την ε, Επίτροπο που προσπάθησε να, προ, προσπαθεί να προχωρήσει την αναμόρφωση αυτή πριν λήξει το τωρινή θητεία. θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ε, και η έκθεση που θα γίνει σε τρία χρόνια να δει πώς ε, λειτουργεί, πώς η διαδικασία. Επίσης εξετάζεται η εισαγωγή νέων τεχνολογιών που θα γίνει με διαβούλευση των ενδιαφερμένων μερών και η προοπτική αξιολόγηση της εφαρμογής. Νομίζω ότι δημιουργεί θεσπίζεται σαφώς με ενόψη της νέας κοινής ελευθερικής ε, πολιτικής. Είναι όλα αυτά θέματα που θεωρώ πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστενσεν, όλα Κρίστενσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για πολύ καιρό χρειάστηκε ε, μία ε, πλήρης αναθεώρηση των ε, κανονισμών ελέγχου και των τεχνικών κανόνων και για την κοινή αλληλευτική πολιτική πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό αποτελεί μεγάλο άχθος για τους αλληλείς όλα μετρώνται, ζυγίζονται και ελέγχονται, αλλά αυτό δεν δημιουργεί πιο βιώσιμη αλία, περισσότερη γραφειοκρατία μόνο. Φυσικά χρειαζόμαστε κοινού κανόνε για να πατάξουμε την απάτη, όμω ε, μέσω τη ε, επιστήμη και τη τεχνολογία. μπορούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε πιο αποτελεσματικά. Πρέπει να συμμορφωθούμε με τι υποχρεώσει στη νέα αλλιευτική πολιτική. Ε, χρειαζόμαστε καλό πλαίσιο για την αλία. Είναι ο μόνος τρόπο για να επιτύχουμε του στόχου μα με τη νέα πολιτική αρχίσουμε λοιπόν τη δουλειά με νέα κοινά, απλά μέτρα ελέγχου που θα οδηγούν σε υγιή ανταγωνισμό και αλία. Ευχαριστώ την συγκήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Έχουμε τώρα κάποια... Ε, τη διαδικασία Κατσδιάη έχουμε δύο ε, αιτήματα. Η κυρία έχει το λόγο. <laughs> u svakom slučaju Ευχαριστώ. Είναι σαφές πως ο κανονισμός αυτός πρέπει να αλλάξει. Η μη, δεν θα υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση. Πρέπει να έχουμε έναν κατάλληλο νομικό έλεγχο. Ταυτόχρονα σύμφωνο με τους συναδέλφους που είπαν ότι η πολιτική αυτή δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα των χωρών μας, της Κροατίας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Προφανώς η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Κάθε χώρα πρέπει να μπορεί να αναπτύξει την δική της αλληλευτική πολιτική. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να κάνουμε τις σχετικές προσπάθειες. Ε, υπάρχουν επιπρόσθετοι πόροι, Κρίμα θα ήταν να μην τους ε, χρησιμοποιήσουμε. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θέλω να εκφράσω την αμφιβολία, τις αμφιβολίες μου ως προς το ότι το Κοινοβούλιο αυτό μπορεί να ελέγξει την υλοποίηση της κοινή ελευτικής πολιτικής εφόσον δεν έχει στη διάθεσή του επαρκείς επιτροπές και εργαλεία για να το κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Σπίκολα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Η αλλαγή από το παλιό σύστημα επιτροπολογίας στο νέο απαιτεί αλλαγή των διαδικασιών λήψης απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φέτος η πολιτική αυτή θα αξιολογηθεί μαζί με τις Διαδικασίε και μεθόδους ελέγχου, τόσο ώστε να ευθυγραμμιστεί με τι ανάγκε τη κοινή ελεκτική πολιτική Πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της τα κατάλληλα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατόπι για εκτελεστικές πράξει και που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των αλλιέων και θα λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένε πρακτικές κρατών μελών. Γι' αυτό υποστηρίζω την, ε, τον έλεγχο ανά τρία έτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τις τελευταίες παρατηρήσεις ε, της Κομισιόν, κύριε Επίτροπος. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Είναι προφανές ότι θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που ήδη είπα, ότι όλες οι παρατηρήσεις και οι ανησυχίες θα ακουστούν, αλλά Φυσικά σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου ε, θα είναι σε προεξέχουσα θέση όπως κατανοείτε. Νομίζω λοιπόν ότι ο διάδοχός μου θα είναι έτοιμος να έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο με μια καλή πρόταση λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις σας. Αλλά επίσης ε, όσον αφορά στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού ε, θα ακολουθηθεί η προτιμόμενη μέθοδος. Κάποια ε, λίγα σχόλια αν μπορώ κύριε Πρόεδρε μόνο. Πρώτον, για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τα ετοιμάσει όλα ώστε να δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη σωστή εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Και γι' αυτό η πρότασή μας ε, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο περιλαμβάνει ένα μεγάλο ποσό το οποίο είναι ε, ακριβώς ταγμένο για αυτή την πολιτική ε, βάση ε, επιστημονικών στοιχείων. Αυτά τα αναφέρατε και κάποιοι από εσάς. Αυτό έχει ως στόχο να δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να έχουν τις δικές τους τεχνικές και να εφαρμόσουν με τον δικό τους τρόπο τους, κανόνες, τους εφαρμοστικούς κανόνες αυτού του κανονισμού. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη διαδικασία περιφερειοποίησης στην ε, μεταρρύθμισή μας, έτσι ώστε ε, τα κράτη-μέλη με βάση την ε, θαλάσσια λεκάνη να μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικά μέτρα, τα οποία θα είναι κατάλληλα για την κατάστασή τους. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια. Αυτό που λέω είναι ότι έχουμε το πλαίσιο για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο μέλλον. Μετά για τα χρήματα. Φυσικά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα αποφασίσουν για το συμβιβασμό ε, μεταξύ των τριών οργάνων. Ε, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπή σχετικά με το εργαλείο χρηματοδότησης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να προκαταβάλω τις συζητήσει εδώ και τις αποφάσεις στο Κοινοβούλιο. Αυτό που θέλω όμως να υπογραμμίσω είναι ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Οι αλληλείς μα χρειάζονται αυτά τα χρήματα, δεν είναι για μα. Οι τα χρειάζονται, επομένως Παροτρύνω το Κοινοβούλιο, κανένα έκκληση και σε όλους ε, να επιταχύνουν τη διαδικασία έτσι ώστε να έχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται ε, μια γνωμοδότηση για να μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουμε με τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για τους αλείς και τη βιομηχανία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την κυρία Τομά και τους Κιώδης για την πολύ καλή εργασία τους σε αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία ε, Επίτροπο. Τελευταία η, η κυρία Τομά.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 Euh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα του συναδέλφου μου. Θα ήθελα να πω στον κύριο Ρόμεβα ή μάλλον να προσπαθήσω να τον καθιχάσω παρότι αποχώρησε στο μεταξύ, ότι σε σχέση με τον κανονισμό για του ελέγχου, αυτό που κάνουμε εμεί είναι να απαντάμε σε μία και μόνο ερώτηση Πώ γίνεται η εφαρμογή με πράξεις κατεξουσιοδότηση ή με εκτελεστικέ πράξει. Να πω επίση στον κύριο Φερέιρα ότι αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στι παράκτιε κοινότητε ε, είναι ένα αίσθημα που δεν αιτιολογείται πάντοτε ότι σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο ε, ο κανονισμός για τους ελέγχους. Λοιπόν, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι με τους οποίους συμφωνώ. Ε, δυστυχώς, Επίτροπε, βλέπω ότι είμαστε ακόμη σε ένα ομιχλώδες τοπίο ως προς την αναθεώρηση. Μας λέτε ότι αυτό που χρειάζονται οι αλληλείς είναι κανόνες που εφαρμόζονται, μα για να εφαρμοστούν πρέπει να είναι γνωστές, ε, γνωστοί οι ε, συνεκτικοί και να μην αλλάζουν αλλάζουν κάθε μέρα, διότι όπως και σας είπα ε, ε, υπάρχει πρόβλημα με τη συλλογή δεδομένων, με τις απορρίψεις. Ε, το 2015 λοιπόν ε, υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει κορεσμός και απόγνωση από πλευράς τους και τα θύματα πάλι θα είναι οι αλληλείς. Ελπίζω λοιπόν για την αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισής μας και κυρίως της εφαρμογής του κανονισμού για τους ελέγχους, ελπίζω όπως σωστά είπατε ότι θα λάβετε διόντως υπόψη τις δικές μας παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Κλείνει η συζήτηση. Αύριο στις 12 είναι η ψηφοφορία. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, στην κοινή συζήτηση για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού.